αλλαγών σε ονόματα αντιπροσωπιών κοινοβουλευτικών από πλευράς ε, EFTD και δύο υποψηφιότητες. αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, ε, στο τέλος της συνεδρίασης θα θεωρούν εγκεκριθέντα όλα αυτά. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε